Ε, εγκριθεί ο διορισμός τους αν δεν διατυπωθούν ε, αντιρρήσεις πριν από το τέλος της σημερινής συνεδρίας. Τελευταία ανακοίνωση, ήθελα να σας ανακοινώσω ότι οι συμπρόεδροι θα υπογράψουν ε, μαζί με τον πρόεδρο του Συμβουλίου έξι νομοθετικές πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 74 του κανονισμού του Κοινοβουλίου. Ε, οι τίτλοι των νομοθετικών αυτών πράξεων θα δημοσιευτούν στα πρακτικά αυτής της συνόδου. Περνάμε τώρα στην ημερήσια διάταξη.